Dear colleagues, good afternoon. Αγαπητοί συνάδελφοι, χαίρετε. Although we are not really numerous. Παρά το γεγονός ότι δεν είμαστε πάρα πολύ πολλοί άριθμοι, νομίζω ότι μπορούμε να αρχίσουμε. As usually, we begin by adopting our... Ως ήθιστε, πρώτο θέμα είναι η έγκριση της ημερήσιας διάταξης θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι τα σημεία 6, 13, 17 και 19 αναβάλλονται. Κύριε Λεμπρετό, κάτι ακούω που δεν είναι γαλλικά ε, στα ακουστικά μου, είναι πρόβλημα μετάφραση υπάρχει. κάτι σε τσέχικα νομίζω είναι. C'est obligatoire le Oui, oui, je, je... Τα τσέχικα είναι υποχρεωτική γλώσσα. Ναι, ομολογώ ότι δεν τα κατέχω πάνω, ακόμα. So, uh, do we have French now? Τώρα ακούτε γαλλικά. Τώρα εντάξει, ναι. So, once again, um, adoption of age. Έγκριση λοιπόν της ημερήσιας διάταξης, στα σημεία 6, 7, 13 και 19 αναβάλλονται. Διαφωνεί κανείς? Όχι από ό,τι βλέπω. Εγκρίνεται ούτως ημερήσια διάταξη. Σημείο 2, ανακοινώσεις του Προέδρου. Θα ήθελα μόνο να σας θυμίσω ότι αύριο θα χρειαστείτε τις ε, κάρτες ψηφοφορίας σας, διότι ψηφίζουμε. Για να μην σας πω και σήμερα. Item number Σημείο 3. Έγκριση των πρακτικών. Εάν δεν έχετε αντιρρήσεις που θα υποβάλλετε μέχρι το τέλος της συνεδρίασης θα θεωρηθούν εγκεκριμένα τα πρακτικά της 22ης και 23ης Μαρτίου 2017. Και τώρα συνεχίζουμε το σημείο 4. Ακρόαση των επιλεγμένων υποψηφίων για τη θέση του Προέδρου του Δευτέρου Τμήματος Προσφυγών του Γραφείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Πνευματική Ιδιοκτησία. Yeah. Όπως γνωρίζετε, όπως ναι, προβλέπει ο αντίστοιχος κανονισμός, η συμμετοχή μας συμμετέχει στην επιλογή των υποψηφίων για τη θέση του Προέδρου του Δευτέρου Τμήματος Προσφυγών του EUIPO, η οποία θέση χειρεύει. Σήμερα θα ακούσουμε τους τρεις υποψηφίους που έχουν επιλεγεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Φυσικά χωριστά τον καθένα. Θα αρχίσουμε τον πρώτο υποψήφιο που είναι ο κ. Φολιάχ. Ε, ε, Καλωσορίσατε ορίσατε. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε σήμερα ενώπιόν μας. Θα έχετε την ευκαιρία να μιλήσετε στην Επιτροπή μας σε 10 λεπτά περίπου. και θα ακολουθήσουν άλλα δέκα λεπτά για ερωτήσεις και απαντήσεις. Αν συμφωνείτε. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρίες και κύριοι. Είναι χαρά μου που βρίσκομαι σήμερα εδώ. Η δήλωσή μου θα είναι κάπως διαφορετική από αυτό που είχα αρχικά σκεφτεί να κάνω και αυτό γιατί είναι, είναι τρεις υποψήφοι και μόνο δύο εθνικότητες που εκπροσωπούνται εδώ. Ε, ένας Γερμανός και δύο Γάλλοι. Και για να μην ε, χαλάσω την ευκαιρία του συνυποψηφίου μου, εγώ αποφάσισα να αποσύρω τη δική μου υποψηφιότητα για να αφήσω το πεδίο ελεύθερο για τον συνάδελφο, όμως ε, θα εκμεταλλευτώ την ευκαιρία για να σας πω πώς βλέπω την δουλειά ε, αυτή στον οργανισμό πνευματικής ιδιοκτησίας και στόχος μου είναι να σας δώσω κάποιες απόψεις για το τι θα ήθελα να επιτύχω ίσως στο μέλλον και με ποιο τρόπο. Σύντομα, δύο λόγια για μένα. Τα πέντε πρώτα χρόνια της επαγγελματικής μου εμπειρίας ε, εργάστηκα σε ένα νομικό γραφείο, εκπροσωπώντας ε, πελάτες, βοηθώντας εταιρείες, καθώς και μεμονωμένους επιχειρηματίες να προστατέψουν τις επενδύσεις τους. Ε, το 2001 συνεργάζομαι σε αυτό το γραφείο. Εργάστηκα για δύο χρόνια στο τμήμα σχεδιασμού μετά από την έγκριση του σχετικού κανονισμού από την Ένωση για τον ε, σχεδιασμό και μετά είχα την ευκαιρία να εργαστώ στην ε, νομική υπηρεσία. 14 χρόνια λοιπόν έχω εργαστεί συνολικά εκεί, περασπίζοντας ε, στηρίζοντας το εφε της διαδικασίες έφεσης σε πάνω από 500 υποθέσεις. Εδώ και πάνω από τρία χρόνια ορίστηκα ως αρχηγός αυτής της ομάδας διευθέτησης ε, ε, διαφορών. Έχουμε 14 ε, δικηγόρους και έχουμε περίπου 400 υποθέσεις ετησίως. Ε, είμαι δηλαδή επικεφαλής αυτής της ομάδας. Στην αρχή, ε, καταρχάς χειρίζομαι τις δικές μου υποθέσεις, έπειτα δίνω κατευθυντήριες γραμμές στους συναδέλφους και εποπτεύω τη δική τους εργασία ώστε να εξασφαλίσω ότι η θέση που κρατάμε ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου είναι σύμμορφη προς τις πρακτικές του γραφείο μας. Και από την εμπειρία μου στην ε, ιδιωτική αυτή πρακτική αλλά και στην διοίκηση έχω αποκομίσει κάποια διδάγματα και ήθελα να σας τα εξηγήσω και σίγουρα αυτά θα ανοίξουν το δρόμο για τις συστάσεις που θα είχα να δώσω σε οποιοδήποτε υποψήφιο για την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού ε, Πνευματικής Ιδιοκτησία. Καταρχάς, μια απόφαση δεν είναι καλή μόνο αν είναι νομικό ορθή. Είναι καλή και, είναι, και γίνεται αντιληπτή ως καλή από τους αποδέχτες της, εάν η απόφαση αυτή αντικατοπτρίζει την ε, ε, γνώση και την συνειδητοποίηση των οικονομικών της επιπτώσεων. Άρα λοιπόν ο επικεφαλής θα πρέπει να γνωρίζει την ε, επιχειρηματική πραγματικότητα πέρα από τα νομικά ε, επιχειρήματα. Αυτό είναι πολύ βασικό για να μπορεί κανείς να λάβει αποφάσεις ε, έχοντας γνώση της, του πλαισίου και του οικονομικού περιβάλλοντος, της οικονομικής κατάστασης. Δεύτερο δίδαγμα που έχω αποκομίσει είναι ότι ένα σημαντικός άξονας είναι επίσης ότι θα πρέπει ο πρόεδρος του οργανισμού είναι να εξασφαλίζει ότι οι, φυστάμενοι του ε, εργάζονται στο έπακρο των δυνατοτήτων τους. Ασκείται πίεση, αλλά αυτό θα πρέπει να γίνεται εις βάρος των, αποφάσεων του Συμβουλίου. Και καθώς είναι ανεξάρτητο, νομίζω πως αυτό είναι πολύ σημαντικό, το να είναι κανείς ανεξάρτητος δεν σημαίνει πως δεν είναι υπόλογος ε, και υπεύθυνο για τις αποφάσεις που λαμβάνει. Άρα λοιπόν ο πρόεδρος του οργανισμού θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται είναι ρεαλιστικές και όχι δογματικές. Κάτι άλλο που αφορά την ποιότητα των αποφάσεων είναι ότι αυτές οι αποφάσεις θα πρέπει να λαμβάνονται με βάση την αξία της κάθε υπόθεσης και να μην ακολουθούνται διαδικαστικές ε, ε, διαδικαστικοί οδοί ώστε ε, να λαμβάνονται οι αποφάσεις. Όποτε είναι δυνατόν αυτό, σημαίνει ηλική δικαιοσύνη στην ουσία, επίτευξη της ηλικής δικαιοσύνης που είναι σημαντική γιατί οι ισχύοντες κανόνες ε, δεν μπορούν να γίνουν δεκτοί όταν αυτό σημαίνει πολλαπλασιασμό αφέσεων, επανάληψη ενεργειών και εν τέλει ε, περί τα κόστη τα οποία φέρουν οι χρήστες του συστήματός μας. Τρίτο δίδαγμα που αποκόμισε οποιοδήποτε αποτέλεσμα επιτυγχάνεται από τον πρόεδρο του Συμβουλίου θα είναι αποτέλεσμα μιας ομαδικής εργασίας. Ο πρόεδρος θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να πείσει τους υπόλοιπους, αλλά και να πιστεί από τους υπόλοιπους. Ο πρόεδρος θα πρέπει να έχει την δυνατότητα να διευρύνει τις γνώσεις του αλλά και, να τις, και τον ενθουσιασμό του και να το μοιραστεί με τα μέλη της ομάδας. Οπότε ο πρόεδρος θα πρέπει όχι μόνο να διευρύνει τις δικές του δεξιότητες, αλλά και αυτές των ανθρώπων με τους οποίους συνεργάζεται. Και αυτό είναι επίσης παράγον κλειδί για να επιτύχει κανείς αποτελεσματική και αποδοτική ομαδική εργασία. Τέταρτο και τελευταίο δίδαγμα που έχω αποκομίσει είναι ότι ομαδική εργασία σημαίνει συνεργασία και με άλλες ομάδες και σε αυτή την περίπτωση με άλλα, συνεργασία με άλλα συμβούλια ε, ώστε συλλογικά αυτά να μπορούν να ακολουθούν συγκεκριμένη γραμμή και ε, νομολογία ούτως για την πρακτική που ακολουθεί το γραφείο μας. Αυτά είναι τα διδάγματα που έχω αποκομίσει με κατόπιν 20 ετούς ε, επαγγελματική εμπειρίας και αυτή θα ήταν η δήλωση που θα είχα κάνει ίσως θα την κάνω και μια άλλη φορά ως υποψήφιος πρόεδρος. και πάντοτε θα έχω στο μυαλό μου ότι μια αυτοχρηματοδοτούμενη, ένας αυτοχρηματοδοτούμενος οργανισμός όπως αυτό το γραφείο εργάζεται ε, με και για ιδιώτες. Αυτό είναι σημαντικό να το έχει κανείς υπόψη του, γι' αυτό έτσι εξασφαλίζει καλύτερη αποδοχή από τους παραλήπτες, τους αποδέκτους των αποφάσεων και έπειτα περιορίζεται και ο αριθμός των εφέσεων ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Ένα άλλο στοιχείο είναι ότι οι πόροι του γραφείου θα πρέπει να ε, αξιοποιούνται στο μέγιστο βαθμό ώστε να ε, λαμβάνονται αποφάσεις που βασίζονται στην ηλική δικαιοσύνη. Όλες οι προσπάθειες θα πρέπει να έχουν στόχο τη διεύρυνση την προσωπικές και επαγγελματικέ δεξιότητες των μελών του Συμβουλίου με καθολικό τρόπο ξεκινώντας από τους νομικούς συμβούλους τα μέλη του Συμβουλίου αλλά και το διοικητικό μηχανισμό, ώστε όλοι να θεωρούν ότι είναι μέλη μια ομάδα και να προσπαθούν συλλογικά να επιτύχουν αποτελέσματα και να συστήνουν ομολογία. Αυτό είναι ο καταλληλότερος τρόπος με τον οποίο θα μπορέσει να εξυπηρετήσει το ε, Συμβούλιο αυτό τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ πολύ. Οπότε καταλάβαμε ότι αποσύρατε την υποψηφιότητά σας. Σωστά καταλάβαμε. Ναι, θα αποσύρω την υποψηφιότητά μου, ναι. Δεν είχα ακόμη το χρόνο να το πράξω, γιατί όπως σας είπα είχα μόλις ε, μία συζήτηση με τον ε, ε, τον άλλο Γάλλο υποψήφιο, γιατί και τελικά αποφασίσαμε από κοινού ναι, το κατάλαβα, το κατάλαβα, αλλά από διαδικαστική απόψη εξακολουθείτε να είστε υποψήφιο. Ναι, αυτό ανέφερα και στην εισήγησή μου, ότι με χρυσό του να αποσύρω την αιτησή μου, ε, παραμένω υποψήφιο. Ναι. Μάλιστα. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι? Ε, I do not see any in that. Δεν βλέπω να ενδιαφέρεται κανείς να ρωτήσει κάτι, εφόσον δεν υπάρχουν ερωτήσεις ε, για σας λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν σκοπεύετε να παραμείνετε υποψήφιος. Σας ευχαριστώ ωστόσο που ήρθατε. Χαίρετε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι χαίρετε. This is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 Uh, Η κυρία Μελγκάρ, είναι δεύτερη υποψήφια. Καλώς ορίσατε στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Θα θέλαμε να σας δώσουμε το λόγο για 10 λεπτά περίπου για να μας ε, κάνετε την εισήγησή σας και 10 λεπτά στη συνέχεια θα έχουμε ερωτήσεις και απαντήσεις. Και Μπορείτε να μιλήσετε οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιθυμείτε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα σας, αξιότιμοι βουλευτές. Θα μιλήσω πρώτα ισπανικά, στη συνέχεια γαλλικά, στα ιταλικά, γερμανικά και τέλος αγγλικά. Ονομάζομαι Μαρία Βερχίνια Μελκάρ, γεννήθηκα πριν από 57 χρόνια σε μια μικρή πόλη της Ουρουγουάης, στην ε, Μίνας. Εκεί πήγα στο δημοτικό και στο γυμνάσιο, σε ένα γυμνάσιο σε Ιταλίδες καλόγριες και ταυτόχρονα μάθαινα αγγλικά στην Αμερικανική Αλιάνς και γαλλικά στην Αλιάνς Φρανσές. Από μικρή ήθελα να γίνω δικαστής και αναγκάστηκα να εγκαταλείψω τη χώρα μου γιατί τότε η Ουρουγουάη ε, υπέφερε ε, από μια στρατιωτική χούντα και αποφάσισα να σπουδάσω στη Γαλλία. Έφτασα στο Παρίσι στην ηλικία των 17 ετών και ε, γράφτηκα σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια, σε μια από τις καλύτερες σχολές νομικής, νομικής ασάς, ε, όπου σπούδασα νομικά και εγκληματολογία στο Γαλλικό Εγκληματολογικό Ινστιτούτο. Μετά τις σπουδές μου επέτυχα στον Εθνικό Διαγωνισμό για το Δικαστικό Σώμα και έγινα πάρεδρος ο Ζουστής το 1982. Μετά από μια διετία ως αντιεισαγγελέας στο Πρωτοδικείο των Βερσαλιών, υπηρέτησα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης σε σχέση με τη διεθνή συνεργασία σε θέματα ε, δίωξης καταστολής και ποινικού δικαίου. Το 1991 επελέγει για να γίνω ε, Γάλλη ρίδα εμπειρογνώμονα στην ε, υπηρεσία, την αντίστοιχη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην νομική υπηρεσία για την εσωτερική αγορά και την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων. Στην αρχή εκπροσωπούσα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, στο ΔΕΚ τότε, για τα προδικαστικά ερωτήματα και το τότε πρωτοδικείο. Επίσης, ήμουν αρμόδι ε, σε θέματα παραβιάσεων κατά των κρατών μελών και το ε, Γενικό Δικαστικό Συμβούλιο. Και τότε άρχισαν να με ενδιαφέρουν τα θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας και βιομηχανικής ιδιοκτησίας από τη σκοπιά όμως ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων και της εσωτερικής αγοράς. την τελευταία χρονιά μου ως Εθνική Απεσπασμένη Εμπειρογνώμων τη πέρασα στη Γενική Διεύθυνση που τότε ονομαζόταν Βιομηχανία, Γενική Διεύθυνση 3 και ήμουν αρμόδια για τις χημικές ουσίες. Ε, τότε είχα προετοιμάσει και ένα διαγωνισμό για να γίνω υπάλληλο Ευρωπαϊκή Επιτροπή, νομομαθή. Επέτυχα στο διαγωνισμό αυτό και λίγο πριν αναλάβω στι Βρυξέλλε έμαθα ε, ότι το νεοσύστατο γραφείο ε, εναρμόνιση τη εσωτερικής Αγορά στο Αλικάντε έψαχνε νομικούς και κατέθεσα την υποψηφιότητά μου, οπότε και επελέγει το Δεκέμβριο του 1994. Άρχισα λοιπόν τη σταδιοδρομία μου στο γραφείο αυτό που τότε ονομαζόταν ε, Σημάτων ε, και Σχεδίων και Μοντέλων τον Ιανουάριο του 1995 στην νομική υπηρεσία πρώτα και μετά στη Διεύθυνση Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων και στη συνέχεια ως επιθεωρήτρια ε, για τα σήματα, δηλαδή για τις αντιρρήσεις και τις ακυρώσεις. Το 2005 επελέγει ε, ως βασική διευθύντρια της νομικής υπηρεσίας ε, του Γραφείου τεχνιών στο Μόναχο, γιατί ήθελα να ασχοληθώ και με ε, μια άλλη πτυχή της πνευματικής ιδιοκτησίας. Τότε είχα αναλάβει θέματα για μια πενταετία θεσμικού χαρακτήρα, να εκπροσωπώ το θεσμό αυτό στον διοικητικό δικαστήριο του ILO και για μια πενταετία ήμουν επικεφαλή 45 νομομαθών από διάφορες χώρες ε, με έδρα την Ολλανδία και τη Γερμανία. Και διαχειριζόμουν και ένα προπολογισμό περίπου 500.000 ευρώ. Επέστρεψα στο Αλικάντε στις αρχές του 2010 και αμέσως ε, ορίστηκα νομικός σε μια υπηρεσία που αφορούσε τις ε, διενέξεις στο δικαστήριο. Δηλαδή, εκπροσωπούσα το τμήμα προσφυγών ε, του γραφείου για πάνω από τέσσερα χρόνια και την 1η Σεπτεμβρίου 2015 έγινα μέλος του 5ου τμήματος προσφυγών του γραφείου και είμαι πανευτυχής εκεί ε, μόνη μου ή με τους συναδέλφους μου χειρίζομαι φακέλους ε, και προσφυγές στα γαλλικά, αγγλικά, ισπανικά και πορτογαλικά. Εκεί εργαζόμαστε και στα Ιταλικά. Συνεπώς οφείλω να παίρνω αποφάσεις στα Ιταλικά ε, σε συνεννόηση και συμφωνία με τους συναδέλφους μου. Επιπλέον, ε, ε, το τμήμα προσφυγών είναι αρμόδιο για προσφυγές και διαδικασίε στα γερμανικά και επιφορτίζονται με την διεκπαιρέωση αυτών οι γερμανόφωνοι συνάδελφοι. Γι' αυτό και πολλές αποφάσεις συντάσσονται στα γερμανικά. Τα γερμανικά είναι η δεύτερη σημαντικότερη γλώσσα εργασίας ε, στο τμήμα προσφυγών. Στο παρελθόν Absolviert. έχω συμμετάσχει σε διάφορα μαθήματα γερμανικών και εξακολουθώ να μετακπαιδεύομαι και σήμερα στη γλώσσα αυτή. Το, τα τμήματα προσφυγών είναι τμήμα της δομής του γραφείου. Συνεργαζόμαστε σε εργαστή συνεργασία και αυτούς είναι από τους στρατηγικούς μας στόχους. Οι αποφάσεις που λαμβάνουμε εγγράφονται στις γραμμές δράσης και συγκεκριμένα στον στόχο 1, να βελτιώνεται η επιχειρησιακή ετοιμότητα και στο στόχο 2 για συστήματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Επίσης και στη γραμμή 5 για να ενισχυθούν οι ποιοτικέ υπηρεσίες με κέντρο τον πελάτη. Και στη ε, γραμμή δράση 6 ενίσχυση του συστήματος πνευματικής ιδιοκτησίας. Προσωπικά πιστεύω ότι μπορούμε ακόμα περισσότερο να ενισχύσουμε την ποιότητα των αποφάσεών μας. Για παράδειγμα μπορούμε να μειώσουμε τους χρόνους που χρειάζονται για να βγάλουμε μια απόφαση. Οχτώ μήνες έχουμε για να εκδώσουμε αποφάσεις και είμαι πεπισμένη ότι αυτό μπορεί να μειωθεί και να φτάσει το εξάμεινο, για παράδειγμα. Αυτό μπορεί να γίνει με τη χρήση εργαλείων που μας βοηθούν να είμαστε πιο αποτελεσματικοί και να εργαζόμαστε ταχύτερα. Είμαι όμως πεπισμένη ότι αυτό που χρειαζόμαστε είναι να βρισκόμαστε πιο κοντά στους χρήστες μας. Γνωρίζετε ότι ο στρατηγικός στόχος του γραφείου για την επόμενη πενταετία είναι ε, να είμαστε ένας οργανισμός ε, ε, εστιασμένος στο χρήστη και είμαι πεπισμένος είναι ότι μπορούμε να προχωρήσουμε προς την κατεύθυνση αυτή. Αυξάνοντας τις ακροματικές διαδικασίες όπου να προσφέρουμε διαμεσολάβηση ή συνδιαλλαγή. Γιατί δεν είναι πάντα μια επίσημη και τυπική λύση ε, της ε, διένεξης ή ε, ενδεδειγμένη. Επίσης, μπορούμε να βελτιώσουμε και την ποιότητα των αποφάσεων στην ουσία, γιατί έχουμε ένα ποσοστό το οποίο ακυρώνει το δικαστήριο των αποφάσεών μας, για παράδειγμα για λόγους διαδικαστικούς. Βέβαια, γύρω στο 85% επιβεβαιώνονται οι αποφάσεις μας, αλλά είμαι βεβαισμένη ότι μπορούμε αυτό να το βελτιώσουμε έτσι ε, περαιτέρω. Έχω την αίσθηση ότι η εμπειρία μου, η ενέργεια μου και η δέσμευσή μου για καλύτερα αποτελέσματα και ποιοτικά και ποσοτικά και χρονικά και εγκύτητα στους χρήστες με καθιστούν ε, κατάλληλη υποψήφια για τη θέση του Προέδρου ε, του Δευτέρου Τμήματος Προσφυγών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία μου. Και τώρα έχει έρθει η ώρα των ερωτήσεων και των απαντήσεων. Ποιος ζητεί το λόγο. Άντερσον. Thank you. I have uh, Ευχαριστώ πολύ. Έχω τέσσερις ερωτήσεις, αλλά θα περιοριστώ σε δύο μόνο ερωτήσεις για να μην σας πάρω όλο το χρόνο. Καταρχήν, θέλω να σας ευχαριστήσω για τις εντυπωσιακές γλωσσικές σας γνώσεις. Θα ήθελα να αναφερθώ σε μία απόφαση που λήφθη το 2015 για την ε, έγκριση ενός ε, σήματος ως κοινοτικού σήματος. Ήταν αρκετά αντιφατική αυτή η απόφαση, διότι αφορούσε ένα γνωστό λογοτεχνικό έργο. Η απόφαση του Συμβουλίου ε, Προσφυγών ακύρωσε την ε, προηγούμενη απόφαση που αρνεί την ε, διεθνή προστασία γιατί δεν πληρούνταν οι κατάλληλες προϋποθέσεις. Και στο Βέλγιο το εφετείο πάλι το 2013 είχε αρνηθεί αυτή την δυνατότητα. Οι, ε, τα πνευματικά δικαιώματα είχαν ε, λήξει το 2016, επομένως θα έπρεπε τώρα να είναι ανοιχτά ε, και δημόσια. Αν δεν υπάρχουν πλέον πνευματικά δικαιώματα γιατί έχουν λήξει. Αυτό το οποίο ζητεί το από το Γραφείο Πνευματικής Ιδιοκτησίας ήταν η καλύτερη προστασία των περιουσιακών στοιχείων αλλά και της πρόσβασης του κοινού στο λογοτεχνικό έργο αφετέρου αν θέλετε να το σχολιάσετε. Και έχω και μια δεύτερη ερώτηση πιο σύντομη. Η ευρωπαϊκή νομοθεσία που εφαρμόζει τη συνθήκη του Μαρακέ είναι το θέμα της δεύτερης ερώτησης. Για καλύτερη πρόσβαση σε βιβλία για τυφλούς. Αυτό θα βοηθήσει βιβλιοθήκες στην Ευρώπη να διαθέτουν αντίτυπα στο κοινό. Συνεχίζονται οι διαδικασίες των τριμερών διαπραγματεύσεων και θέλω να σας ρωτήσω πώς σκοπεύει το Γραφείο Διανοητικής ε, Ιδιοκτησίας να βοηθήσει σε αυτή τη διαδικασία. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Κάουφμαν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε κυρία Μέλγκα. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίασή σας. Μια ερώτηση έχω να σας κάνω. όσον αφορά την ανεξαρτησία που απαιτείται στο αξίωμα αυτό. προβλέπετε στον κανονισμό ότι ο πρόεδρος ε, του Συμβουλίου Προσφυγών και τα μέλη θα πρέπει να είναι ανεξάρτητα και να μην δεσμεύονται κατά κανένα τρόπο για τη λήψη αποφάσεων κατά τις ε, δραστηριότητές τους. Θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς ε, σκοπεύετε να εγγυηθείτε ότι θα υπάρξει στην πράξη τέτοια ανεξαρτησία. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Φως. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ έχω μία ερώτηση, ίσως και δύο ερωτήσεις. Πρώτον, το Συμβούλιο Προσφυγών έχει μια συγκεκριμένη διαδικασία και θα ήθελα να σας ρωτήσω ποια είναι η δική σας θέση όσον αφορά το δικαίωμα της ακρόασης και πώς θα υπάρχει εγγύηση της ανεξαρτησίας. Ήδη σας τέθηκε η πρώτη ερώτηση σχετικά με την ανεξαρτησία του Συμβουλίου Προσφυγών η πιο σημαντική σας επαγγελματική εμπειρία την οποία προσφέρετε στο νέο σας αξίωμα για το οποίο είστε υποψήφιο ποια είναι. Πρόεδρος, έχετε το λόγο κυρία Μέλγκαρ για να απαντήσετε στις ερωτήσεις που σας ετέθησαν. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ενδιαφέρουσες οι ερωτήσεις αυτές. Όσον αφορά την πρώτη ερώτηση για το σήμα Αν Φρανκ, μπορώ να σας δώσω και μια προσωπική απάντηση και μια θεσμική απάντηση. Υπήρξε πολύ μεγάλη συζήτηση και πολλές διαφορές στο γραφείο σχετικά με την απόφαση αυτή. Εγώ προσωπικά σοκαρίστηκα γιατί πιστεύω ότι δεν θα έπρεπε να δεχόμαστε ένα σήμα για βιβλία, διότι ο κανονισμός ε, λέει ότι δεν θα πρέπει να εξετάζουμε ποιος υποβάλλει αίτηση για σήμα. Από την άλλη πλευρά, ο νομοθέτης λέγει ότι υπάρχουν σήματα, ονόματα και λογότυπα που πρέπει να είναι ελεύθερα, να, μπορεί να τα χρησιμοποιεί ε, ο πολίτης στην καθημερινότητα. Προσωπικά, εγώ θα είχα δώσει αρνητική απάντηση σε ένα σήμα για βιβλία. Πιστεύω ότι αυτό δεν συνάδει προς την φιλοσοφία του νομοθέτου. Όμως, τονίζω ότι ήταν πολύ μεγάλες οι συζητήσεις και οι διαφορές σε ολόκληρη την Ευρώπη για το θέμα αυτό. Και τώρα και στο μέλλον εταιρείες θα προσπαθούν να αποκτήσουν μονοπόλιο, γιατί το σήμα ουσιαστικά αυτό τους δίνει, ένα αποκλειστικό δικαίωμα. Κάποιες εταιρείε φτάνουν πρώτες, υποβάλλουν την αίτηση και μπορούν να έχουν ένα μονοπόλιο επάπειρον, αν κάθε δέκα χρόνια το ανανεώνουν. Μια πρόσφατη υπόθεση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ασχολήθηκε με ένα ε, διαφορετικό θέμα για ένα πολύ γνωστό βιβλίο στη Γερμανία, το Winnie Two μέσα, στο μέσα στον επόμενο μήνα νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θα μας δώσει πολύ ξεκάθαρες οδηγίες για τέτοιου είδους σήματα ούτω ώστε να μπορέσουμε και εμείς να τροποποιήσουμε τις οδηγίες μας και να εξηγούμε γιατί τέτοιου είδους σήματα δεν μπορούν να γίνονται δεκτά. Και κάποιες εθνικές αρχές κρατών μελών αντιμετώπισαν παρόμοια ζητήματα και έλαβαν διαφορετικές αποφάσεις από το γραφείο. Σας έδωσα τώρα την προσωπική μου θέση. Είμαι πεπισμένη ότι στο μέλλον δεν θα προκύπτουν τόσο αντιφατικά ζητήματα γιατί θα δει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σαφέστερες κατευθύνσεις. Τώρα όσον αφορά τη συνθήκη του Μαρακές και την υποστήριξη που μπορεί να παρέχεται. Ένας από τους στόχους του στρατηγικού σχεδίου τώρα είναι να ενισχυθεί η γνώση σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα είτε στο παραδοσιακό μας αντικείμενο, δηλαδή σήματα και σχέδια, ή και πνευματική ιδιοκτησία και δικαιώματα ευρεσιτεχνίας. Η Ακαδημία που είναι ένα από τα τμήματα του γραφείου που ασχολείται με την ανάπτυξη, προσφέρει online σεμινάρια και μια πλατφόρμα online, διαδικτυακή και πάλι, όπου μπορούν να συζητούνται θέματα πέραν των σημάτων και των σχεδίων. Το σύστημα αυτό λειτουργεί για τα θέματα που αποτελούν το βασικό μας κορμό μέχρι τώρα, αλλά προγραμματίζουμε και επέκταση. Έχουμε κάποια σχέδια για το Μητρό των Ορφανών Έργων, κάποια παρακολούθηση μέσω του παρατηρητηρίου. Πιστεύω δηλαδή ότι όλο και περισσότερο θα μπορούμε να προσφέρουμε βοήθεια στην ανάπτυξη τεχνογνωσίας. Περνώ τώρα στην επόμενη ερώτηση σχετικά με την ανεξαρτησία του Συμβουλίου Προσφυγών. Η ανεξαρτησία μας θεσπίζεται από τον κανονισμό. Και πέραν της, πέραν της θεσμικής ανεξαρτησίας είναι και θέμα προσωπικού χαρακτήρα. Ε, από το παρελθόν μου ως δικαστικού, με την εκπαίδευσή μου στην Εθνική Σχολή Δικαστών και με την εμπειρία μου ως εισαγγελέα, που δεν είναι καθόλου προφανές δεν είναι καθόλου εύκολο να μπορεί κανείς ε, να αναλάβει μια τέτοια θέση αν δεν έχει εγγυημένη ανεξαρτησία. Πιστεύω ότι είναι θέμα προσωπικότητας και χαρακτήρα η εγγύηση της ανεξαρτησίας. Όταν στόχος μας είναι το κράτος δικαίου και όταν ε, είμαστε και υπό τον έλεγχο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, είναι σχετικά πιο εύκολο να θεωρούμε ότι είναι εγγυημένη η ανεξαρτησία. Εγώ ε, μπορώ να προσφέρω 35 χρόνια εμπειρίας σε ποικίλου διεθνείς οργανισμούς και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτός το παρελθόν μου από το δικαστικό τομέα νομίζω με έχει προετοιμάσει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τη θέση αυτή και για την διασφάλιση της ανεξαρτησίας του Συμβουλίου. Στο γραφείο και τώρα, αλλά και σίγουρα και στο μέλλον, επικρατεί μια πολύ καλή ατμόσφαιρα όσον αφορά τη θεσμική διακυβέρνηση και μας σέβονται όλοι. Δεν είμαι καθόλου απεσιόδοξη λοιπόν για το μέλλον και το κατά πόσο θα έχουμε ανεξαρτησία στο μέλλον. Τα Συμβούλια Προσφυγών επιτελούν εξαιρετικό έργο το οποίο το έχει αναγνωρίσει και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Και αυτό οφείλεται στο ότι έχουμε ενστερνιστεί αυτή την ανεξαρτησία την οποία και εκφράζουμε. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας. Δεν βλέπω να υπάρχει κάποια επιπλέον ερώτηση. Σας ευχαριστώ που ήσασταν σήμερα εδώ και παρακαλώ αν θέλετε να περάσετε έξω τώρα. Uh, Κύριε Στούρμαν, καλώς ήρθατε στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Έχετε 10 λεπτά για την αρχική σας δήλωση. Θα ακολουθήσουν ερωτήσεις από τους βουλευτές και θα έχουμε άλλα 10 λεπτά για ερωτήσεις και απαντήσεις συνολικά. Έχετε το λόγο. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Πριν αρχίσω, θα ήθελα ε, να εκφράσω ε, το σεβασμό μου για τον κύριο Φωλιά και την εκτίμησή μου που απεσύρθη από, την υποψηφιότητά μου. Θα ήταν καλός υποψήφιος και θέλω να πω ότι τον ε, εκτιμώ ιδιαίτερος. Κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και αγαπητά μέλη της Επιτροπής ε, Τζούρι, σας ευχαριστώ που με καλέσατε σε αυτή την ακρόαση. Για μένα είναι μεγάλη τιμή το ότι βρίσκομαι σήμερα ενώπιόν σας ως υποψήφιος για τη θέση του Προέδρου του Δευτέρου Τμήματος Προσφυγών ε, της, ε, του Γραφείου δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, ε, υποψήφιο ε, που έλαβε τις, την πλειοψηφία των ψήφων των κρατών μελών για τον κατάλογο υποψηφίων που είχε καταρτήσει το Συμβούλιο Διοίκηση του EU IPO. Και είναι μεγάλη τιμή για μένα να σας παρουσιάσω το όραμά μου για το ρόλο του Προέδρου. Όταν ήμουν παιδάκι, πήγαινα συχνά με τον πατέρα μου σε επισκέψει που έκανε σε πελάτες του το Σαββατοκύριακο. Και όταν ήμασταν στο αυτοκίνητο με τον πατέρα μου, μου έλεγε πάντοτε «Γεια μου, πρέπει να είμαστε διαφανείς και συνεπείς σε ό,τι κάνουμε και να ακούμε προσεκτικά ό,τι μας λένε οι πελάτες μας και να ακούμε όλες τις ανησυχίες τους». Έκτοτε, πάντοτε αυτό αποτέλεσε ένα βαθύτερο κίνητρο και στην προσωπική και στην επαγγελματική μου ζωή. Από την αρχή της καριέρας μου στο EU IPO, φιλοδοξία μου ήταν να συνεισφέρω στο να γίνει η δημόσια διοίκηση πιο διαφανής, περισσότερο συνεπής και περισσότερο αποτελεσματική στην υπηρεσία των πολιτών. Και γι' αυτό το όραμά μου για το Συμβούλιο Προσφυγών είναι το να αποτελέσει ένα βασικό τμήμα αριστείας στο, σύστημα του ευρωπαϊκού, στο ευρωπαϊκό σύστημα ε, πνευματικής ιδιοκτησίας. Αν εκλεγώ ο πρόεδρος, ε, θα προσπαθήσω να ε, συνεισφέρω για την εκπλήρωση αυτού του οράματος με τις ιδέες και τις εμπειρίες μου και θα εστιαστώ σε τρεις τομείς. Πρώτον, συνέπεια και συνοχή των ε, διαδικασιών και των αποφάσεων ε, σχετικά με τις προσφυγές. Δεύτερον, αποτελεσματική επίλυση διαφορών πνευματικής ιδιοκτησίας. Και τρίτον, ενισχυμένη συνεργασία με τους εθνικούς φορείς προσφυγών. Όσον αφορά τη συνέπεια και τη συνοχή, τα Συμβούλια Προσφυγών παίζουν βασικό ρόλο στη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Σημάτων και Σχεδίων και ε, δημιουργούν το υπόβαθρο για την ε, πρωτοβάθμια διαδικασία του EUIPO και ε, χρησιμεύουν ως σημεία αναφοράς για τα εθνικά δικαστήρια, τα εθνικά όργανα προσφυγών και τα εθνικά γραφεία πνευματικής ιδιοκτησίας. Ως εκ τούτου η συνέπεια και η συνοχή είναι απαρέγκλητες. Επίσης, από την έναρξη των εργασιών των Συμβουλίων το 1996, αυξάνονται οι προσφυγές και οι περισσότερο χρησιμοποιούμενες γλώσσες είναι τα αγγλικά και τα γερμανικά. Μόνο 10% των αποφάσεων ε, είναι αντικείμενο προσφυγών το δικαστήριο, το οποίο στη συνέχεια επιβεβαιώνει το 85% των αποφάσεων των Συμβουλίων Προσφυγών. Και αυτό αποδεικνύει ότι είναι πολύ υψηλή η ποιότητα εργασιών των Συμβουλίων. Αλλά βέβαια δεν μπορούμε να επαναπευθούμε στι δάφνε μα. Πρέπει συνεχώ στα Συμβούλια Προσφυγών να βελτιώνουμε τι εργασίε μα για να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε στι αυξανόμενε ανάγκε των χρηστών. Και αυτή είναι μια τεράστια πρόκληση και απαιτεί όχι μόνο νομικέ γνώσει, αλλά και δεξιότητε σε θέματα διοίκηση και ηγετικέ ικανότητε. Εγώ έχω τι ικανότητε για να ανταποκριθώ στην πρόκληση αυτή, διότι έχω νομική εμπειρία, όπως επίσης και εμπειρία σε θέματα ηγεσία και διοίκηση. Σπούδασα νομική στη Γερμανία και στην Ισπανία με επίκεντρο το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και έχω και μεταπτυχιακό δίπλωμα στο, στην πνευματική ιδιοκτησία. 15 ε, χρόνια εργάστηκα ως ε, δικηγόρος σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας, πρώτον ε, στον ιδιωτικό τομέα και στη συνέχεια στο EUIPO, στο πρωτοβάθμιο επίπεδο, στο νομικό τμήμα και στα συμβούλια προσφυγών, χρησιμοποιώντα καθημερινά την αγγλική, γερμανική, ισπανική και γαλλική γλώσσα. Είμαι επίση μέλο του Συμβουλίου Προσφυγών ε, του Γραφείου Φοιτικών Ποικιλιών στην Ανζέ. Αυτέ οι θέσει μου έχουν δώσει τη δυνατότητα να βλέπω τα δικαιώματα πνευματική διοκτησία από πολλέ διαφορετικέ ε, γωνίε. Εκτό τη νομική μου εμπειρία έχω και εμπειρία σε θέματα διοίκηση και ηγετικών θέσεων. Ήμουν επικεφαλής ε, του επιχειρησιακού τομέα της EUIPO και τώρα είμαι επικεφαλής της ομάδας του Συμβουλίου Προσφυγών και Program Manager και ως επικεφαλής του κύκλου γνώσεων σε διαδικασίες προσφυγών ε, καθοδήγησα τις προσπάθειες των Συμβουλίων Προσφυγών ε, σε μια προσπάθεια εναρμόνισης των ε, διαδικασιών προσφυγών υπέρ των χρηστών μας. Αυτές οι εμπειρίες δείχνουν τις δεξιότητές μου και ως νομικού και ως ατόμου με ηγετικές ικανότητες με τη δυνατότητα να εμπνέω και να δίνω κίνητρα σε ομάδες από πολλούς τομείς και πολλές ιδιότητες και διαφορετικά πολιτισμικά πλαίσια. Και τέλος έχω ανοιχτό πνεύμα και έχω την ενέργεια και το ενδιαφέρον και το ζήλο για νέες προκλήσεις. Όσον αφορά την αποτελεσματική επίλυση διαφορών πνευματικής ιδιοκτησίας, είμαι πεπισμένος ότι μέσα στις προκλήσεις της εποχής μας πρέπει να δείξουμε ότι η διοίκηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ανοιχτή, γρήγορη και διαφανής και ότι ενδιαφέρεται για τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των πολιτών και των εταιριών. Παραδείγματο χάρη μπορεί η ίδια ε, πλευρά να είναι ε, ο, ο ίδιος διάδικος να βρίσκεται σε διαδικασίες ταυτόχρονα στα Συμβούλια Προσφυγών και ενώπιον εθνικών δικαστηρίων και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θα πρέπει σε τέτοιες ε, περιπτώσεις να χρησιμοποιούμε ε, μηχανισμούς με τους οποίους θα μπορούν οι χρήστες να έχουν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην επίλυση των διαφορών τους πρόσφατα σε μία σύστασή σας προς την Επιτροπή για τα κοινά ελάχιστα πρότυπα πολιτικής δικονομίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εσείς αντιμετωπίσατε το θέμα αυτό. Και η δική μου άποψη για το πώς θα αντιμετωπίζετε ένα τέτοιο θέμα είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει μία σωστή διοίκηση όπου ο εισηγητής θα πρέπει μαζί με τους διαδίκους να αποφασίζει για τον πιο αποτελεσματικό μηχανισμό επίλυσης ε, διαφορών. Η απόφαση των συμβουλίων ή ε, μεσολάβηση ή συνδιαλλαγή. Ο χρήστης είναι στο επίκεντρο αυτών των προσπαθειών και θα πρέπει να δίνουμε στον χρήστη τις δυνατότητες να αντιμετωπίζεται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο η διαφορά τους ε, χωρίς περιττό κόστος και καθυστερήσεις. Για το λόγο αυτό έπαιξα βασικό ρόλο στη δημιουργία της ε, Υπηρεσίας ε, Μεσολάβησης των Συμβουλίων Προσφυγών, όπου εμπνευστήκαμε από την Οδηγία Μεσολάβησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου του 2008. Θέλουμε να δείξουμε στους χρήστες ότι τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι όχι μόνο ενεργά στο νομοθετικό πεδίο, αλλά ότι επίσης εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Ένωση το πνεύμα της Οδηγίας της Μεσολάβησης ο πρόεδρος παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια αυτό. Ο πρόεδρος ή η πρόεδρος θα πρέπει να καθοδηγεί και να διευκολύνει το αποτελεσματικό σύστημα επίλυση διαφορών. Θεωρώ ότι είμαι κατάλληλο άτομο για να διασφαλίσω την ομαλή λειτουργία μιας, ενός τέτοιου συστήματος ε, διαχείρισης υποθέσεων στο Συμβούλιο Προσφυγών. Έχω λάβει πολλές φορές αποφάσεις, είμαι πεπειραμένος σε τέτοια θέματα και έχω εργαστεί στα Συμβούλια Προσφυγών για πολλά χρόνια, έχοντας συντάξει εκατοντάδες αποφάσεις και είμαι και ο πιο πεπειραμένος ε, μεσολαβητής του EUIPO. Τέλος, ε, όσον αφορά την ενίσχυση της συνεργασίας με τα εθνικά όργανα προσφυγών, τα Συμβούλια Προσφυγών θα πρέπει όχι μόνο να εστιάζουν την προσοχή τους στη λήψη αποφάσεων και στην αποτελεσματική επίλυση διαφορών πνευματικής ιδιοκτησίας, αλλά θα πρέπει να ε, μπορούν να μοιράζονται τις γνώσεις και την εμπειρία τους σε διάλογο με άλλους εταίρους όπως είναι τα εθνικά δικαστήρια, τα εθνικά όργανα προσφυγών και τα εθνικά γραφεία πνευματικής ιδιοκτησίας. Ο Ευρωπαίος νομοθέτης ε, έχει δείξει σαφώς ότι θα πρέπει να συνυπάρχουν το ευρωπαϊκό και τα εθνικά συστήματα σημάτων και σχεδίων. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να διδασκόμεθα ημένα από τους ΔΕ και θα πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ τι κάνουν οι εθνικοί εταίροι μας, ιδίως όσον αφορά το EUIPO και τα γραφεία προσφυγών, τα οποία υπάρχουν τα τελευταία 20 χρόνια, ενώ τα εθνικά συστήματα πνευματικής ιδιοκτησίας υπάρχουν πάνω από 100 χρόνια. Επομένως, αν εκλεγώ πρόεδρος, θα προσπαθήσω να εξασφαλίσω καλύτερη συνεργασία μεταξύ των Συμβουλίων Προσφυγών του EUIPO και των Εθνικών Οργάνων Προσφυγών, των Εθνικών Γραφείων Πνευματικής Ιδιοκτησίας, ούτω ώστε να καθορίσουμε τις βέλτιστες πρακτικές και για να μπορούμε να διδασκόμεθα ημένα από τους ΔΕ. Εν κατακλείδη, με βάση αυτές τις ε, ιδέες, εάν εκλεγώ πρόεδρος, θα συνεισφέρω για να γίνει πιο αποτελεσματικό και συνεπές το Συμβούλιο Προσφυγών, ώστε να, μπω, να μπορώ μια μέρα να πω στην κόρη μου ότι έχω ολοκληρώσει την αποστολή μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας και περιμένω τις ερωτήσεις σας. Σας ευχαριστούμε. Υπάρχουν Έχετε ερωτήσεις ε, προς τον υποψήφιο. Ο κύριος Φως. Ευχαριστώ κύριε Θα Σας ευχαριστούμε για την παρουσίασή σας. Αναφέρατε και τη μεσολάβηση. και η Επιτροπή Νομικών ε, Υποθέσεων ε, το Μάρτιο ασχολήθηκε με μια οδηγία σχετικά με τη μεσολάβηση. Τι έχετε κάνει εσείς για τη μεσολάβηση και πώς βλέπετε το ρόλο της μεσολάβησης στο μέλλον. Αυτό είναι το πρώτο μέρος της ερωτησής μου. Και το δεύτερο μέρος της ερωτησής μου θα είναι πιο σύντομο. Ε, θα ήθελα να σας ρωτήσω τι βαρύτητα έχουν οι γλώσσες ε, ε, στην ενασχόληση των τμήματων προσφυγών με τις διάφορες υποθέσεις. Για να βελτιώσουμε τη συνέπεια και τη συνοχή των αποφάσεων, ίσως θα πρέπει να έχετε και υποστήριξη από σύγχρονες τεχνολογίες. Ο κύριος Άντερσον, σας ευχαριστώ. Έχω δύο ερωτήσεις που θέλω να ε, ρωτήσω τον υποψήφιο. Πρώτη, αναφέρεται σε μια απόφαση που ελήφθη το 2015 από την ε, EUIPO για έγκριση εμπορικού σήματος για τον όρεο Dairy Frank ως κοινοτικό εμπορικό σήμα. Είναι αρκετά επίμαχη. Ε, γιατί ε, αυτό το σήμα αντιπροσωπεύει ευρωπαϊκή ε, ευρωπαϊκή λογοτεχνική δημιουργία. Όμως παλιότερα είχε απορριφθεί η σχετική αίτηση, είχε γίνει ωστόσο έφεση στο Βέλγιο. Τώρα, αυτό το σήμα εξέπνευσε το, 2, η Ιανουαρίου 2016 και σύμφωνα με τους σχετικούς κανόνες θα πρέπει πλέον να ανήκει, να είναι πλέον δημόσιο ε, αγαθό. Όμως αυτή η απόφαση είναι αντίθετη με το νομοθεσία περί ε, πνευματικής ιδιοκτησίας και το αίτημα, η έφεση μάλλον κατετέθη από ε, την ε, ε, εταιρεία. Δεν ξέρω, θέλω να μου πείτε αν εσείς θα μπορέσετε να τραβήξετε ξεκάθαρη γραμμή ανάμεσα στα συμφέροντα ιδιωτών για την προστασία των δικών τους περιουσιακών στοιχείων είτε είναι πνευματικά είτε όχι και την άλλη πλευρά το δημόσιο συμφέρον. Τώρα, σε σχέση με την, Αμερικανική, την συνθήκη του Μαρακές για την πρόσβαση των τυφλών σε βιβλία. Ε, ε, ο προβληματισμός αφορά πώς θα μπορέσουν να βοηθηθούν οι, αρμόδιοι οργανισμοί όπως οι βιβλιοθήκες να προσφέρουν ε, πνευματικά έργα σε ανθρώπους με προβλήματα όρασης. Πώς λοιπόν το γραφείο θα μπορέσει να βοηθήσει αυτούς τους αρμόδιους οργανισμούς, τους συγκεκριμένου οργανισμούς, αυτό το έργο κατά τη γνώμη σας. Ευχαριστώ. Αυτές είναι οι ερωτήσεις και τώρα έχετε ε, τη δυνατότητα να απαντήσετε. Σας ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις. Αν μου επιτρέπετε να απαντήσω στην πρώτη. Να απαντήσω στα γερμανικά. Το θέμα της διαμεσολάβησης πρώτα. Το 1999 σπούδασα ε, διαμεσολάβηση και μάλιστα ήταν η πρώτη φορά που προτινόταν αυτός ο κύκλος σπουδών και έχω εργαστεί ως ε, διαμεσολαβητής δικηγόρος και συνεισέφερα πραγματικά σημαντικά ε, στο δικό μας σύστημα ε, προσφυγών και μάλιστα έχει και επιστοποίηση ISO αυτή η διαδικασία στη Γερμανία και διάβασα μια σύντομη ε, παρουσίαση ε, που είναι πολύ ενδιαφέρουσα, μου επιτρέπετε ε, να σας τα αναφέρω. Είναι εξασφάλιση της ποιότητας, πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο. Συμφωνούμε πολύ με τη σύστασή σας. Θα πρέπει να είναι εγγυημένη η ποιότητα. Στέλνουμε επιστολή και μάλιστα κάνουμε έρευνα ικανοποίηση του πελάτη. Για να δούμε αν μπορούμε να βελτιώσουμε την ποιότητα. Και τρεις φορές το χρόνο έχουμε μια προσωμείωση, μια άσκηση προσωμείωσης διαμεσολάβησης για να βελτιωνόμαστε. Για αυτό για το πώς λειτουργεί η υπηρεσία μετά. Ε, ένα πολύ σημαντικό συμπέρασμα που είδα στην έκθεση αυτή ήταν ότι στιγματίζεται το γεγονός ότι δεν υπάρχει ούτε πληροφόρηση ούτε γνώση επαρκή στα κράτη-μέλη για την ύπαρξη καν αυτή της διαδικασίας. Πραγματικά η συστέση αυτή είναι πάρα πολύ σωστή. Θα πρέπει όλο και περισσότερο να δούμε με ποιον τρόπο ε, μπορούμε να προβάλλουμε και να διαφημίσουμε στον κόσμο την μεσολάβηση ιδιαίτερα τα πλεονεκτήματα για τους πολίτες και τις εταιρείες. Εμείς το κάνουμε αυτό στα Τμήματα Προσφυγών ο εισηγητής κάστοτε αναλύει την περίπτωση και αποφασίζει και κοιτάζει αν είναι δυνατόν να ε, προτείνουμε τη μεσολάβηση Δεν είναι πάντα αυτό δυνατό σε όλες τις διαδικασίες και στη συνέχεια ε, προτείνουμε στα μέρη τη διαδικασία αυτή. Εγώ ενθαρρύνω τον κόσμο προς την κατεύθυνση αυτή και είναι σημαντικό γιατί και η ιδέα της έκθεσης είναι αυτή ότι θα πρέπει εμείς να βγούμε προς τον κόσμο και να τους εξηγούμε ποια είναι τα πλεονεκτήματα, οι ιδιαιτερότητες, το όφελος. Τότε ο κόσμος το βλέπει πιο ανοιχτά και ιδιαίτερα οι δικηγόροι και ρωτούν, α ναι, έχει νόημα, ποια είναι τα πλεονεκτήματα, θα πρέπει εμείς να βγούμε προς τον κόσμο να κάνουμε περισσότερα για να προβληθεί και να γίνει γνωστή η διαδικασία αυτή της διαμεσολάβησης. Το κάνουμε σε ε, άρθρα που γράφουμε, σε διασκέψεις, σε, σε διοργανώσεις ένα θέμα που έχει να κάνει το μέλλον και έχει να κάνει και με το τελευταίο σας ερώτημα. Η διαμεσολάβηση εξοδικαστική στο μέλλον πραγματικά ε, ε, είναι σημαντική γιατί ε, φέρει ένα βάρος από τη δικαιοσύνη και φέρει και τους ανθρώπους πιο κοντά. Τώρα αποφασίστηκε μια δικαστική μεταρρύθμιση, το άρθρο 137α ετέθησε εισήγη πέρυσι για να συσταθεί μια ε, αντίστοιχη υπηρεσία πρωτόδικα. Γιατί ε, τώρα η διαμεσολάβηση υπάρχει ε, στη δεύτερη φάση, στη φάση της προσφυγής, αλλά όχι στη βάση της εξέτασης των διενέξεων και των διαφορών. Για τη δεύτερη ερώτηση, για τις γλώσσες. Εργαζόμαστε και στις 23 γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή οι εταιρείε και φυσικά πρόσωπα, εκτός από τα νομικά πρόσωπα, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για ονομασία, για σήμα και στις 23 ε, γλώσσες, αλλά 46% ε, πέρσι ήταν αγγλικά, 70% ε, ήταν γερμανικά, 7, 8 ισπανικά και άλλες γλώσσες. Το ίδιο ισχύει και για το τμήμα προσφυγιών. Από τις 2.884 ε, περιπτώσεις, 64% ήταν ε, αγγλικά, 23% γερμανικά και 5% των διαδικασιών ισπανικά και 3% ε, γαλλικά. Καταλαβαίνετε ποιες είναι οι γλώσσες οι συχνότερες, κυρίως αγγλικά και γερμανικά κατά δεύτερο λόγο. Και στο δεύτερο τμήμα πρόσφυγων λόγω της σύνθεσης σήμερα δεν μπορεί να εξετάσει διαδικασία, στην ακροαματική διαδικασία στα γερμανικά. Δηλαδή μοιράζονται υποθέσεις στα υπόλοιπα τμήματα. Ακριβώς επειδή υπάρχει τέτοιος φόρτος και τόσες πολλές ε, ε, περιπτώσεις στα γερμανικά και υποθέσεις, καλό θα ήταν και το δεύτερο τμήμα να μπορεί να τις εξετάζει στα γερμανικά. Για τη συνοχή και τη συνεκτικότητα, για το διαδίκτυο και πόσες σύγχρονες τεχνολογίες μπορούν να ε, χρησιμοποιηθούν. Ενδιαφέρουσα πτυχή αυτή και σημαντική. Ίσως να γνωρίζετε ότι ο εκτελεστικός μας διευθυντής, Αντώνιο Καμπίνος, από την αρχή, από την πρώτη του θητεία, εργάστηκε για ένα στρατηγικό σχέδιο του 2015 μέχρι 2020 και επέμεινε πάρα πολύ στη χρήση νέων τεχνολογιών ακριβώς για να είμαστε πιο συνεκτικοί, πιο συνεπείς και πιο αποτελεσματικοί για τους πολίτες και τις ε, εταιρείε να καταφεύγουν σε εμά για τις ε, υποθέσεις τους. Ε, όλες οι υποθέσεις, σχεδόν όλες, μπορεί να γίνουν και επιγραμμικά. Και πριν από τρεις εβδομάδες έχουμε εισαγάγει μια νέα εφαρμογή μας για επιγραμμικές καταγγελίες και παράπονα. Εγώ είχα την αρμοδιότητα και το συντονισμό αυτού του νέου λογισμικού. 30.000 αποφάσεις έχουμε λάβει τα τελευταία 20 χρόνια στο Τμήμα προσφυγών και από την άλλη έχουμε και εκατοντάδες ή μάλλον χιλιάδες αποφάσεις του Πρωτοδικίου του Δικαστηρίου ε- της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μην μιλήσουμε για την εθνική δικαιοσύνη και οπότε είναι πολύ σημαντικό να προωθήσουμε την ε, τεχνολογία και τις υποθέσεις στο διαδίκτυο. Επανέρχομαι τώρα στα αγγλικά, απαντώ στην ερώτησή σας, αν σας κατάλαβα καλά. Ε, αναφερθήκατε ε, στο σήμα Άννα Φρανκ. Με κάθε σεβασμό, αυτό είναι μια απόφαση του τέταρτου τμήματος προσφυγών του 2015 είναι ενδιαφέρον το ερώτημά σας. Ε, βέβαια το αυτή τη στιγμή είναι λίγο δύσκολο να απαντήσω γιατί είμαι υπάλληλο του οργανισμού αυτού και δεν μπορώ να σχολιάσω υπερβολικά αυτή την απόφαση. Πάντως, από πλευράς copyright και προστασίας έχει σημασία. Αυτό που είπατε, πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε μια ισορροπία ανάμεσα σε ένα ιδιωτικό συμφέρον και εκείνον που δημιούργησε το έργο και το δημόσιο συμφέρον. Πολύ σημαντικό. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι φυσικά πρέπει να βρεθεί μια ισορροπία. Θα πρέπει να ακολουθήσουμε την νομολογία του ε, Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης τώρα μάλλον και του Γενικού Δικαστηρίου. Χωρίς αποκλεισμούς και λαμβάνοντα υπόψη την ισορροπία των ενδιαφερομένων μερών. Προς τα εκεί θα πρέπει να κινηθούμε και να βεβαιωθούμε ότι εφαρμόζει την ομολογία Η συγκεκριμένη περίπτωση εκεί εντάσσεται. Και να με ειλικρινής, το δεύτερο τμήμα της ερώτησή σα δεν το πολύ κατάλαβα. Για τους τυφλούς. Ποια ήταν η ερώτηση. Στο μικρόφωνο παρακαλούμε. Να την επαναλάβω. Πώς προτίθεται το γραφείο να βοηθήσει τη διάδοση των βιβλίων για τυφλούς. Α, πώς μπορούμε εμείς να βοηθήσουμε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης και στη διάδοση των έργων. Μπορούμε να υποστηρίξουμε, φαντάζομαι. Θα πρέπει να σκεπτόμαστε δημιουργικά. Αλλά αν υπάρχει απόφαση που λέει ότι κάποια έργα θα πρέπει να είναι προσφάσιμα και σε ανθρώπους με προβλήματα όρεσης ή τυφλούς, θα πρέπει εμείς να δημιουργήσουμε ενδεχομένω τα απαραίτητα εργαλεία για να διευκολυνθεί αυτή η πρόσβαση, η, η διάθεση. Τώρα δεν έχω να σας πω συγκεκριμένα τι αυτό μετάφραση αν υπάρχει όμως απόφαση σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να το κοιτάξουμε φυσικά. Και από εκεί και πέρα βλέποντας και κάνοντας και να αποφασίσουμε πώς μπορούμε να το μεταφέρουμε στην πράξη. Για να διευκολύνουμε την πρόσβαση στα έγγραφα αυτά. Thank you very much for, uh, Σας ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις στα ερωτήματα των ε, μελών και που ήρθατε Σας παρακαλώ όμως τώρα να βγείτε έξω. So, dear colleagues, as you know, it is not our role. Συνάδελφοι, όπως γνωρίζετε, ο ρόλος μας δεν είναι να επιλέξουμε έναν από τους δύο υποψήφιους. Εμείς ε, θα πρέπει να συντάξουμε μία γνωμοδότηση. Έχουμε συμφωνήσει λοιπόν με τη Γραμματεία ότι θα ετοιμάσουν ένα σχέδιο επιστολής και με τους συντονιστές θα το εγκρίνουμε και θα το στείλουμε όπου δει. Ωραία, ευχαριστώ. Να περάσουμε τώρα στο σημείο περθών 5. Εξέταση της γνωμοδότησης σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της συνθήκης όσον αφορά τα εθνικά κοινοβούλια. Και το λόγο έχει ο κύριος Λεμπρετό. Merci, Monsieur le Président. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Προτείνω να εντάξουμε στην πρόταση ψηφίσματος τα εξής. Καταρχάς, διαβάζοντας την ετήσια έκθεση 2015, φαίνεται ότι οι σχέσει ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα Εθνικά Κοινοβούλια παραμελείται σε πολύ μεγάλο βαθμό ο πρωταρχικός ρόλος των Εθνικών Κοινοβουλίων από πλευρά των Κομισιών, για να μην πούμε και ότι υπάρχει μια υποτίμηση της αξίας τους, περιφρόνηση. Αυτό συζητήσαμε και χτες ε, όπου ένας ε, Τσέχος γερουσιαστής είπε ότι οι αιτιολογημένες νομοδοτήσεις των Εθνικών Κοινοβουλίων πολύ σπανίως ακολουθούν το από σχετικές ενέργειες και ότι ακόμα πολλές φορές και η κίτρινη κάρτα δεν λαμβάνεται επαρκώς υπόψη. Τα Εθνικά Κοινοβούλια ωστόσο είναι η, μόνη, η, άμε, η πιο άμεση και νομιμή ε, θεμητή μάλλον εκπροσώπηση της δημοκρατίας στα διάφορα κράτη-μέλη της Ένωσης και εξάλλου η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει αυτό τον καθοριστικό ρόλο, τον εξέχοντα ρόλο μέσω της αρχής της επικορικότητας που θα έπρεπε να προστατεύει τη δράση των Εθνικών Κοινοβουλίων. Και χθε η συζήτηση στην ΑΦΚΟ επιβεβαίωσε το ζήτημα αυτό, καθώς ο ε, διευθυντής του Ινστιτούτου Χάμπλε ε, μάλλον επιβεβαίωσε ότι τα Εθνικά Κοινοβούλια αποτελούν την νομιμότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του να μην γίνονται σεβαστά δεν εμπίπτει στο πνεύμα αυτού του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Θεωρώ επίσης πως η Κομισιόν, αν και υπογραμμίζει τη σημασία ενός εις βάθος διαλόγου, ε, τελικά κρύβεται πίσω από το δικό της μονοπόλιο της νομοθετικής πρωτοβουλίας ώστε τελικά αυτός ο διάλογος να μην ε, φτάσει σε τίποτα το συγκεκριμένο να μην καταλήξει σε τίποτα το συγκεκριμένο και σίγουρα θα πρέπει αυτό να μας απασχολήσει δηλαδή το μονοπόλιο της νομικής πρωτο... νομοθετικής πρωτοβουλίας. Επίσης υπάρχει συστηματική προσφυγή της Κομισιόν στη διαδικασία κατεξουσιοδότησης πράξεων που είναι υποτίθεται η κατεξαίρεση διαδικασία αλλά γίνεται πλέον ε, ε, κατακόρων και το Ίδρυμα Σούμαν δείχνει ότι δύο τρίτα της νομοθεσίας διαπώνται από τέτοιες κατεξοδότηση πράξεων. αυτή τη στιγμή, δηλαδή η Κομισιόν ε, μπαίνει στη θέση του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και νομοθετεί, πράγμα το οποίο είναι πολύ ανησυχητικό. Να υπογραμμίσω τέλο ότι το έγγραφο το οποίο σχολιάστηκε περισσότερο από τα Εθνικά Κοινοβούλια το 2015 είναι ακριβώ το πρόγραμμα εργασία 2015 τη Κομισιόν, πράγμα που επιβεβαιώνει κατά τη γνώμη μου την καθοριστικό και εξέχοντα νομοθετικό ρόλο που έχει η ίδια δώσει στον εαυτό τη η Κομισιόν. Γι' αυτό και καλό την Κομισιόν να σεβαστεί την αρχή τη επικορικότητας και να περιοριστεί μόνο στις δικέ της αρμοδιότητε και αποστολέ. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ο κύριος Βιέφκα ζητά τώρα το λόγο. Bardzo dziękuję panie przewodniczący, σας ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ ευχαριστώ τον συνάδελφο Λεμπρετών για την έκθεσή του για τη γνωμοδότηση αυτή που αφορά το πολύ σημαντικό ρόλο των Εθνικών Κοινοβουλίων στην νομοθετική διαδικασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες είναι ένα θέμα που αρκετά συχνά ε, έρχεται στη συζήτηση γιατί εδώ και χρόνια προσπαθούμε να εμπλέξουμε τα εθνικά ε, κοινοβούλια στην νομοθετική διαδικασία. Εγώ δεν συμφωνώ με τον κύριο Λεμπρετόν όσον αφορά την, τα περισσότερα που καταγγέλει εναντίον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι αλήθεια πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το μονοπόλιο όσον αφορά την νομοθετική πρωτοβουλία, αλλά δεν μπορούμε να ξεχνάμε πως δεν είναι η ίδια η Κομισιόν που από μόνη της ανέλαβε αυτό το μονοπόλιο. Αυτά τα οποία αναφέρετε στην γνωμοδότησή σας οδηγούν σε ένα συμπέρασμα, εάν συμφωνήσουμε μαζί σας. Μόνο μία προοπτική δηλαδή θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε, δηλαδή να τροποποιήσουμε τις συνθήκες. Ο ρόλος των Εθνικών Κοινοβουλίων εντάσσεται στη συνθήκη. Ορίζεται από τη συνθήκη, δεν είναι ελεύθερο πεδίο δράσης ή μη δράσης η αδράνειας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι το μόνο όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει όντως το μονοπόλιο της πρωτοβουλίας και η Κομισιόν δεν νομοθετεί η ίδια. Συμφωνώ λοιπόν ότι γίνονται αρκετέ κατεξοδότητε συμπράξεις, αλλά αυτό είναι σφάλμα της ίδια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να απαντήσουμε έντιμα. Ποιος επιτρέπει στην Επιτροπή να υιοθετεί κατεξοδότηση πράξης. Αυτή η Κομισιόν δεν τις ε, παίρνει τις αποφάσεις μόνη της. Το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο της το επιτρέπουν. Εάν λοιπόν θέλουμε να επιστήσουμε την προσοχή κάποιου σε αυτή την υπόθεση, στον υπερβολικό αριθμό δηλαδή κατεξοδότηση πράξεων, θα πρέπει να επιστήσουμε την προσοχή του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου ε, σε αυτό το γεγονός. Βεβαίως η Κομισιόν μπορεί να έχει την πρωτοβουλία, αλλά εμείς αποφασίζουμε αν η Κομισιόν ή όχι θα, αναλάβει θα έχει τη δυνατότητα. Λέτε έπειτα ότι θα πρέπει να προσέχουμε περισσότερο τον ρόλο των Εθνικών Κοινοβουλίων γιατί είναι τα μόνα δημοκρατικά εκλεγμένα όργανα. Αυτό όμως δεν είναι αλήθεια. Και εμείς ε, είμαστε ε, πρόσωποι της Ευρωπαϊκής Κοινωνίας των Ευρωπαϊκών Λαών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από το 1979 εκλέγεται από άμεσες και καθολικές εκλογές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βεβαίως, όπως και οι κυβερνήσεις στα κράτη-μέλη, δεν εκλέγεται άμεσα Ωστόσο, εσείς ε, θα κατηγορούσατε την κυβέρνησή σας ότι δεν εκλέγεται άμεσα, ενώ αυτό κατηγορείται την Επιτροπή, ότι δεν εκλέγεται άμεσα και ότι μόνο το Ευρωκοινοβούλιο εκλέγεται άμεσα. Έχουμε μία γραμμή συνεργασίας ανάμεσα στα τρία θεσμικά όργανα η Κομισιόν που έχει την πρωτοβουλία και τους δύο συνομοθέτες Συμβούλιο και Κοινοβούλιο. Η εργασία που γίνεται τώρα από την ε, Συνταγματική Επιτροπή θα πρέπει να στηριχτεί από σοβαρές παρεμβάσεις και όχι από ευχολόγια. Να μην πούμε δηλαδή στη Συνταγματική Επιτροπή, απλούστατο, αλλάζουμε τη συνθήκη αλλά πιστεύω πως δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να γίνει κάτι τέτοιο. Θα πρέπει να κάνουμε επικοδομητικές προτάσεις. Ευχαριστώ. Κάποιος άλλος θέλει να πάρει το λόγο. Ο κύριος Άντερσον. Thank you. I have read this uh, Ευχαριστώ. Διάβασα αυτή την πρόταση γνωμοδότησης αλλά δυσκολεύομαι να καταλάβω προς τι μας είναι χρήσιμη για την Συνταγματική Επιτροπή. Επικρίνει την Επιτροπή, ίσως και υπερβολικά, αν μου επιτρέπετε να το εκφράσω έτσι, χωρίς να παρουσιάζει κάποιες εναλλακτικές λύσεις για το τι θα θέλαμε να έχουμε. Νομίζω ότι η Συνταγματική Επιτροπή θα διαμορφώσει μια καλή έκθεση. Και αν εμεί υποβάλουμε μια γνωμοδότηση, καλό θα ήταν να προσπαθούμε να βοηθούμε την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων και αυτή η γνωμοδότηση δεν νομίζω ότι το επιτυχάνει αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Χέγνεχ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομη, αν και θα μπορούσα να μακρηγορήσω. Θέλω απλώς να τονίσω αυτό που είπε ο κύριος Σφιεύκα και ο κύριος Άντερσον. Συμφωνώ απολύτως μαζί τους. Ε, θα ήθελα να πω κάτι όλοι βρισκόμαστε κάπως απομονωμένοι στο ρόλο μας. Εμείς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι βουλευτές στα Εθνικά Κοινοβούλια. Αυτό το οποίο γίνεται στο Αυστριακό Κοινοβούλιο για διευκόλυνση του είναι ότι ε, καλό θα ήταν να μπορούσαν να λαμβάνουν το λόγο οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ολομέλεια του Αυστριακού Κοινοβουλίου. Όταν υπάρχουν δηλαδή ευρωπαϊκά θέματα, να μπορούν να εμφανιστούν οι ε, ομιλητέ στην Ολομέλεια και όχι μόνο σε ειδικέ επιτροπέ. Γιατί όταν συζητούνται πραγματικά τα θέματα και έχουμε πραγματική συζήτηση, όχι μόνο σε μία ώρα συζήτηση για τα ευρωπαϊκά θέματα, να μπορούσαμε να συνεισφέρουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε για την ε, ιδέα αυτή. Μήπως η Επιτροπή θέλει το λόγο. Δεν θέλει το λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σημειώστε λοιπόν ότι η προθεσμία για κατάθεση τροπολογιών είναι η 10η Μαΐου 2017. Κλείνουμε λοιπόν το θέμα αυτό και συνεχίζουμε με το σημείο 7. Εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης για την κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιριών. Η κυρία Ρέγνε είναι η και έχετε το λόγο κυρία Ρέγνε. Ευχαριστώ πολύ. Μόλις έρχομαι από από μια πολύ ενδιαφέρουσα ακρόαση για το ίδιο θέμα στην Επιτροπή Οίκων. Άκουσα δηλαδή ήδη αυτά τα οποία λέγονταν εκεί και πήρα κάποιες ενδιαφέρουσες ιδέες. Θα ήθελα λοιπόν πριν περάσω στην παρουσίαση να σας μεταφέρω κάτι που είπαν οι εκπρόσωποι των μικρομεσαίων επιχειρήσεων γιατί ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η ακρόαση δίπλα οι εκπρόσωποι των μικρομεσαίων επιχειρήσεων γνωρίζουν τι πραγματικά σημαίνει το να πρέπει να αντιμετωπίσουν 28 διαφορετικά φορολογικά συστήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι πολύ μεγάλες εταιρείες δεν υποφέρουν ιδιαίτερως γιατί έχουν τη δομή και έχουν τη δυνατότητα να περάσουν από το ένα νομικό σύστημα και φορολογικό σύστημα στο άλλο. Αλλά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πλήττονται ιδιαίτερως και τις ενδιαφέρει ιδιαίτερως και η κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιριών και η κοινή βάση φορολογίας εταιριών. Παρότι ακούγεται σαν γλωσσοδέτης αυτό το οποίο έχουμε ως τίτλο της γνωμοδότησης αυτής. Πρέπει λοιπόν να έχουμε δικαιοσύνη. Αυτό ενδιαφέρει περισσότερο τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και στη γνωμοδότηση αυτή τονίζω ότι έχουμε δύο προτάσεις το υπόβαθρο το γνωρίζετε, δεν χρειάζεται να το επαναλάβω ούτε για τα έγγραφα του Παναμά, ούτε για τις διάφορες πολιτικές συζητήσεις που έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Είναι απολύτως απαραίτητο σε ένα σύστημα το οποίο είναι παγκοσμοποιημένο και ψηφιακό και με μεγάλη κινητικότητα, να μην ε, βρίσκονται τα κράτη-μέλη ε, πίσω από αυτά τα οποία γίνονται, να μην υπάρχει καθυστέρηση που υπάρχει τώρα. Χρειαζόμαστε και τα δύο αυτά συστήματα, και το CCCTB, Κοινή Ενοποιημένη Βάση Φορολογίας Εταιριών, και την Κοινή Βάση Φορολογίας Εταιριών. Και τα δύο τα χρειαζόμαστε. Είναι πολύ σημαντική η δέσμη αυτών των μέτρων. Δεύτερον, ε, σημαντικό είναι το κατόφλι. Η κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρεών θα πρέπει να είναι υποχρεωτική για όλες τις εταιρείες εκτός από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επανέρχομαι στον ορισμό που έχουμε στην οδηγία για τα λογιστικά. Έχουμε τον ορισμό των μεγάλων επιχειρήσεων και των μικρών επιχειρήσεων Πρέπει να κρατήσουμε αυτή τη διαφοροποίηση και γι' αυτό τόνισα και τη θέση των εκπροσώπων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από την ακρόαση. Τρίτο σημείο είναι το θέμα της καινοτομίας και των επενδύσεων. Γνωρίζουμε ότι χρειαζόμαστε την καινοτομία, χρειαζόμαστε μια Ευρώπη που θα προχωρήσει στο μέλλον και δεν θα είναι απειρχαιωμένη και οι επιχειρήσεις θα πρέπει να επενδύουν τα κέρδη τους στο μέλλον. Η προώθηση της καινοτομίας και των επενδύσεων θα πρέπει να γίνεται μέσω δημοσίων ε, επιχορηγήσεων και όχι μέσω φορολογικών απαλλαγών. Και αυτό το λέω γιατί δεν θέλουμε να έχουμε ένα διάτριτο σύστημα. Συχνά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, έχουμε καλές ιδέες και ένα σημείο δεν προσέχουμε και αυτό γίνεται παραθυράκι για διάφορες εξαιρέσεις και παρεκκλήσεις. Πρέπει λοιπόν να, να μην έχουμε φορολογικές απαλλαγές, αλλά να δίνονται δημόσιες ενισχύσεις για την ε, καινοτομία και τις επενδύσεις. Και εμείς εδώ στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων πρέπει να δείξουμε πνεύμα καινοτομίας σε όλες τις επιτροπές όπου συζητείται αυτό το θέμα, εκεί στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, ε, όπου συζητούνται τα θέματα αυτά επί χρόνια, δεν ε, έχουμε ακόμη μιλήσει για ψηφιακές εταιρείες, γιατί ναι, υπάρχουν όλες αυτές οι επιχειρήσεις όπως η Google και το Facebook και εταιρείε οι οποίες δημιουργούν έσοδα σε ένα κράτος μέλος χωρίς να είναι εγκατεστημένες ε, στο συγκεκριμένο κράτος μέλος, όπως δηλαδή δουλεύει η Amazon και άλλες εταιρείε. Θα πρέπει να θεωρούμε τις ψηφιακές εταιρείε ε, ως εταιρείε που έχουν φορολογική βάση σε αυτή τη χώρα. Είναι μεγάλη πρόκληση γιατί χρειαζόμαστε ένα ορισμό για αυτές τις εταιρείε. Δεν έχουμε τέτοιο ορισμό και τώρα στην Επιτροπή Οίκων συζητήθηκε το θέμα αυτό. Ο κύριος Φέμπερ το ανέφερε το θέμα των σημάτων, το θέμα ε, των ε, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Πάλι μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα όταν οι εταιρείε μεταφέρουν τα κέρδη τους από τη μία χώρα στην άλλη. Ε, ήρθα σε επαφή με το τμήμα ε, μελετών του Κοινοβουλίου και ζήτησα τη γνώμη του σχετικά με ένα τέτοιο ορισμό. Θα έπρεπε να λέμε ότι είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο οικονομικών δραστηριοτήτων που ε, κινητοποιούνται σε πλατφόρμες διαδικτυακές ή κινητές πλατφόρμες μια τέτοια βάση θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε πάνω στην οποία θα πρέπει να χτίσουμε ένα πραγματικό ορισμό. Για μας ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εδώ υπάρχει μια ευκαιρία να δείξουμε πνεύμα καινοτομία και να ορίσουμε τις ψηφιακές επιχειρήσεις. Περιμένω τη συνεργασία με τους συναδέλφους και όδης ε, και ευρωβουλευτές εν γέννη. Ευχαριστώ. Κύριε Φως. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η κυρία Λεγκρίπ είναι σκιώδης εισηγήτρια από πλευράς Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για αυτές τις γνωμοδοτήσεις και ζητεί συγγνώμη για την απουσία της σε αυτή την ανταλλαγή απόψεων. Εξ ονόματός της θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ευγενικά για την παρουσίασή σα και το έργο σας σε όλο αυτό το θέμα. Και η ε, θέλει να αναγνωρίσει τη σημαντική ε, αυτή ε, δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τέτοια μέτρα τα έχουμε συζητήσει εδώ και καιρό στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η έγκριση των προτάσεων αυτό θα σήμαινε ένα μεγάλο βήμα προς μια πιο αποτελεσματική και συνεπή νομοθεσία στην Ευρώπη. Έτσι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορέσει να εντείνει τη μάχη κατά της φοροαποφυγής και να βελτιώσει την εσωτερική αγορά ε, παρέχοντας ε, στις επιχειρήσεις ε, περισσότερη διαφάνεια για το φορολογικό σύστημα της κάθε χώρας ε, και έτσι θα είχαμε περισσότερη διαφάνεια στην οικονομική ζωή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τη σύστασή του αυτή θα ε, καθορίσει τη θέση του και ελπίζουμε τα κράτη-μέλη που έχουν και τον τελικό λόγο για αυτά τα θέματα ε, να ε, ε, συνεργαστούν επικοδομητικά στο Συμβούλιο και να αποδώσει αυτό το σημαντικό εγχείρημα. Η κυρία Λεγκρίπ ακόμα μελετάει την πρόταση της κυρίας Ρέγνερ στο σχέδιο γνωμοδότησής της και προβλέπει στη συνεργασία της μαζί σας για αυτό το σημαντικό θέμα. Ευχαριστώ. I do not see... Δεν βλέπω άλλον κανένα δει το λόγο. Κύριε Τζιγόν. Δύο λόγια μόνο κύριε Πρόεδρε. Ε, συνεχίζοντας ε, από τον προλαλήσαντα, θα ήθελα να πω στην Εύελιν Ρέγνερ ότι φυσικά εμείς συμφωνούμε, δεν λέω ότι η ζωή είναι τέλεια και ο κόσμος θαυμαστός αγγελικά πλασμένος, γιατί θα μας κατηγορήσει ότι είμαστε υπερβολικά ευγενική και καλή μαζί της. Πάντως, εμείς θέλουμε να υπάρχει ενιαία φορολογική βάση στην Ευρώπη και θέλω να καθησυχάσω τον συνάδελφο Λεμπρετό. Τελικά τα κράτη-μέλη έχουν τον τελευταίο λόγο. Μην τρομάζετε, μην ανησυχείτε. Και ακριβώς εμείς μπορούμε να γνωμοδοτήσουμε ε, όσο γίνεται πιο επικοδομητικό τρόπο. Το θέμα της κοινή φορολογικής βάσης είναι ε, κρίσιμο. Γιατί ε, βλέπουμε ότι τα κράτη-μέλη έχουν επιδοθεί σε μια κούρσα ανταγωνισμού και είναι περίεργο να ε, μπορούμε να εξηγούμε ότι για τις υπηρεσίες και τα αγαθά η εσωτερική αγορά λειτουργεί απρόσκοπτα, ενώ έχουμε καθημερινή ε, κούρσα για τα φορολογικά και κόντρα των κρατών μεταξύ τους ένα μικρό ε, θέμα. Εκτός από την έκθεση αναχώρα υπάρχει και ε, το κατόφλι, το όριο 750 εκατομμύρια, 40 εκατομμύρια. 40 εκατομμύρια είναι αν θέλουμε να κάνουμε μια διάκριση ανάμεσα στις μικρές και τις μεγάλες επιχειρήσεις. Το ίδιο θα πρότεινα όπως με την έκθεση ένα χώρο. Να κάνουμε τη διάκριση μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις και να μην έχουμε 750 εκατομμύρια κατόφλι που ε, αφορά μόνο το 10% των εταιριών που δραστηριοποιούνται στην αγορά μας. Ας περάσουμε λοιπόν στα 40 εκατομμύρια που είναι αυτό της οδηγίας για τα λογιστικά θέματα για τις μικρές επιχειρήσεις. Είναι ο αντίστοιχος ορισμός. Ευχαριστώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να λάβει το λόγο. Όχι. Α, θέλει όμως, ναι. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλουμε να εκφράσουμε την υποστήριξή μας και την ευγνωμοσύνη μας για την κοινή φορολογική βάση και την ενοποιημένη ε, φορολογική βάση. Καθώς ορίζουμε τη γενική υποστήριξη ε, των βουλευτών και της εισηγήτριας. Για μας η πρόταση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική με διπλό στόχο. Ο πρώτος είναι η δικαιοσύνη ε, σαφέστατα για να έχουμε ένα σύστημα δίκαιο και ανθεκτικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, φορολογικό, αλλά ταυτόχρονα και ανταγωνιστικό ένα σύστημα φορολογία των επιχειρήσεων που να οδηγεί στην ανάπτυξη και στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης εργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επίσης να είναι συμβατό και στο διεθνές πλαίσιο με τη διεθνή λειτουργία των εταιριών μας για να μπορούν να ανταγωνίζονται ε, άλλες εταιρείε μη ευρωπαϊκές. Εξού και δύο προτάσεις που έχετε σήμερα ε, προς συζήτηση. Επίσης εκτιμούμε το γεγονός ότι εστιάζεται ε, στο στοιχείο της δικαιοσύνης που περιέχει η πρότασή μας, αλλά θα θέλαμε να λαμβάνετε υπόψη και το στοιχείο της ανταγωνιστικότητας, που είναι εξίσου σημαντικό. Νομίζω ότι έχουμε κοινό συμφέρον να προωθήσουμε ένα σύστημα βιώσιμο, ε, δίκαιο, να πληρώνουν τους φόρους που τους αναλογούν ε, με δικαιοσύνη εταιρείε και να μπορούν ταυτόχρονα να ανταγωνίζονται άλλες εταιρείε δίθνως. Σας ευχαριστώ πολύ ε, για το ενδιαφέρον που δείχνετε για το θέμα αυτό και προσβλέπουμε στη μελλοντική μας συνεργασία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν θέλει η συγγετρία να επανέλθει. Όχι. Ωραία. Μπορούμε λοιπόν να κλείσουμε εδώ το θέμα αυτό. Ουσιαστικά το 7 και το 8 συζητήσαμε από κοινού, αν δεν απατώμε. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Προχωρούμε. Σημείο 9. Έχουμε το σχέδιο γνωμοδότησης με θέμα τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχήρωσης των επαγγελμάτων. Και θα δώσουμε και πάλι το λόγο στον κύριο Λευγατό. Τον εισηγητή. Merci, Monsieur le Président. L'Union européenne compte environ 5 5.600 είναι τα επαγγέλματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, που θέλουν κατοχήρωση ειδική. Αυτή, ε, αυτός ο κανονισμός παραμένει ε, προτεραιότητα, μάλλον αρμοδιότητα των κρατών μελών και κάθε ε, κράτος μέλος μπορεί να επιβάλλει όρους ε, ή περιορισμούς στην πρόσβαση στο επάγγελμα αυτό, στην άσκηση του επαγγέλματος, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σήμερα φρονεί ότι δεν υπάρχει ισότητα στην εφαρμογή αυτού και αυτό επηρεάζει ανετικά την παροχή υπηρεσιών, λέει, και την κινητικότητα των επαγγελματιών. Για να διορθώσει αυτή την κατάσταση, προτείνει την οδηγία αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να υπάρχει ένας έλεγχος αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέων νομοθετικών ε, κανόνων για την κατοχήρωση των επαγγελμάτων. Ο εισηγητής σας, ο αποφαινόμενος δηλαδή, δεν συμφωνεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να χρησιμοποιήσει την οδηγία που είναι ε, δεσμευτικό μέτρο. Θα αρκούσε μία σύσταση, κατά τη γνώμη μου, για ελάχιστα κριτήρια για τα κράτη-μέλη ε, που οφείλουν να τα εφαρμόζουν κατά τον έλεγχο της αναλογικότητας. Η Γερμανική Άνω Βουλή επίσης συμφωνεί. Το θέμα αυτό του ελέγχου έχει πολύ λεπτομερή κριτήρια και η πρόταση οδηγίας υπερβαίνει κατά πολύ ε, την νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστήριου υπερβαίνει δηλαδή το στόχο και επιβάλλει ε, στα, σε εθνικές αρχές ε, τον τρόπο με τον οποίο θα κάνουν τον έλεγχό τους και τους δυσκολεύει. Γι' αυτό έχω κάνει κάποιες τροπολογίες που είναι πολύ άριθμες για να τις ε, αναφέρω όλες. Απλώς προσέξτε την τροπολογία παριθμών ένα που θυμίζει την ομολογία του ε, Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκής Ένωσης που θυμίζει την αρμοδιότητα των κρατών για πολλά επαγγελματά όπως είναι το συμβολιογράφο ας πούμε. Ε, η τροπολογία 2 που δίνει κατευθυντήριες γραμμές και όχι κοινή ε, προσέγγιση που είναι πιο διεισδυτική μέθοδος και πιο επιθετική. Η τροπολογία 5 που ε, προβλέπει αντιστροφή του βάρους της απόδειξης. Δηλαδή δεν αναπόκειται πλέον στα κράτη-μέλη να αποδείξουν την αναλογικότητα, αλλά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποδείξει την έλλειψη αναλογικότητας. Εδώ λοιπόν πολύ συγκεκριμένες προτάσεις και επικοδομητικές θα συμφωνήσετε πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Νίμπλα. Ευχαριστώ πολύ κύριε πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ και τον εισηγητή μας για την παρουσίαση των τροπολογιών του και της νομοδότησης. Τρία σχόλια θα ήθελα να κάνω στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ε, συμφωνώ με τον εισηγητή, δεν βλέπω καμία αναγκαιότητα να είναι ε, υποχρεωτικός ο τρόπος του ελέγχου αναλογικότητας για διάφορους λόγους. Καταρχάς πιστεύω ότι ε, το πώς ρυθμίζονται τα επαγγέλματα είναι κράτος των κρατών μελών. Το ακούσαμε και από τον εισηγητή. Και δεν είναι μόνο δική του άποψη, δική μου, ε, πολλών άλλων, αλλά και ε, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που επανειλημμένα έχει πει ότι τα κράτη-μέλη καταρχάς και καταρχήν ορίζουν ποια είναι τα ρυθμισμένα επαγγέλματα. Στη συνέχεια θέλω να πω ότι δεν υπάρχει καν νομική βάση για την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν πρόκειται καν για την αμοιβαία αναγνώριση τίτλων και πιστοποιητικών και πτυχίων. Η νομική βάση που επικαλείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ε, στοιχειοθετεί ούτε δικαιολογεί την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και τρίτον, θέλω να θυμίσω ότι και σε εθνικό επίπεδο αλλά και με την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου αλλά και με την οδηγία για την αναγνώριση των επαγγελμάτων Ξέρουμε τι εστί αναλογικότητα, δεν χρειάζεται να το επαναορίσουμε. Υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια ε, τα οποία έχουν εξηγηθεί και στην οδηγία για την αναγνώριση των επαγγελμάτων, αλλά και με την ομολογία του ΔΕΚ. Οπότε δεν πιστεύω ότι υπάρχει καν ανάγκη να ασχοληθούμε με αυτή την πρόταση και να μπούμε στα χωράφια των αρμοδιοτήτων της, ε, των κρατών μελών και να επέμβουμε. Τέλος, επιτρέψτε μου να κάνω μια γενική παρατήρηση γιατί υποθέτω ότι έχουμε παρόντες εκπροσώπους Ευρωπαϊκής Επιτροπής και για αυτό το θέμα, πάντα όταν προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ρύθμιση επαγγελμάτων, έχω την αίσθηση ότι η αξία της αυτορύθμισης των ελευθέρων επαγγελμάτων ούτε αναγνωρίζεται ούτε εκτιμάται. Γιατί το κάνει αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδώ και χρόνια. ισχυρίζεται ότι δεν συνάδουν αυτά λέει με την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων. Καμία σχέση. Ε, εγώ όλες ε, τις εμπειρίες που έχω ε, με τις οργανώσεις αυτών των επαγγελματιών τις θεωρώ πάρα πολύ θετικές. Φροντίζουν το επάγγελμα, φροντίζουν την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη μετεκπαίδευση και κάνουν εξαιρετική δουλειά οι σύλλογοι των ελευθέρων επαγγελματιών. Για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η καχυποψία και αυτή η δυσπιστία. Μπορεί και να κάνω λάθος, αλλά όταν κάνεις προτάσεις Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι, ότι είναι κατά της αυτορύθμισης των ελευθέρων επαγγελμάτων και δεν συμφωνώ καθόλου, γιατί έχω εμπειρία ετών, πολλών, με τους συλλόγους των επαγγελματιών αυτών. Αντίθετα, με την αυτορύθμιση αφαιρείς και ένα βάρος από το κράτος. Αν δεν το κάνουν οι ίδιοι επαγγελματίες, θα πρέπει να το κάνει το κράτος τον έλεγχο τη ε, ποιότητα. το κατά πόσο αυτό θα ήταν πιο αποτελεσματικό, τολμώ να το αμφισβητήσω. Μεγάλο ερωτηματικό. Εγώ είμαι μέγα οπαδός αυτών των αυτορυθμιζομένων ελευθέρων επαγγελμάτων, του τρόπου με τον οποίο αυτορυθμίζονται. Οπότε θεωρώ και τι προτάσει του εισηγητού μα πολύ καλέ. Αυτά, σύντομα, ω πρώτη ανάλυση. Thank you very much. Uh, Μάλιστα, δεν ζητά κανείς άλλο το λόγο, οπότε ε, να ρωτήσω την Κομισιόν αν θέλει να πάρει το λόγο, να αντιδράσει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εποφελούμε τις διερμηνίες, να μιλήσω κι εγώ γερμανικά. Σας ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον που δείχνετε. Γνωρίζουμε τους προβληματισμούς. Έχουμε ήδη ακούσει τα σχετικά με τα νομικά κοτοχυρωμένα ε, ε, επαγγέλματα. Γνωρίζουμε ε, και τα θέματα επικουρικότητας και αναφέρθηκε και η Γερμανική Άνω σε αυτά τα οποία ακούσαμε. Θα προσπαθήσω να εξηγήσω γιατί εμείς είμαστε της γνώμης ότι περνάμε ε, από το στάδιο της σύστασης στο στάδιο της δεσμευτικής νομικής πράξης. Υπάρχει νομική βάση προς τούτο. Θα είμαι σύντομος, γιατί στην αξιολόγηση επιπτώσεων έχουμε εξηγήσει λεπτομερώς το σκεπτικό μας. Η ιδέα του ότι απαιτείται ένα δεσμευτικό νομικό μέσο για την εξέταση της αναλογικότητας πριν ενός νέου νομικού μέσου είναι σημαντικό κριτήριο. Και αυτή η ιδέα βασίζεται στη βάση της οδηγίας για τα προσόντα που μιλάει για αξιολόγηση και για ανάγκη διαφάνειας Υπάρχουν περίπου 5.700 επαγγέλματα τα οποία θεωρούνται νομικά κατοχυρωμένα. Και προσπαθούμε να έχουμε κάποια αξιολόγηση για να αποδεικνύεται ότι υπάρχει αναλογικότητα για, την, για τα κατοχυρωμένα επαγγέλματα. Έχει γίνει μακρά συζήτηση στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για ε, να βρεθεί η σωστή νομική βάση ώστε να είναι δεσμευτικό αυτό το οποίο προτείνουμε. μετά από ε, πολιετή νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου καταλήξαμε σε αυτό το οποίο προτείνουμε στα κράτη-μέλη και γι' αυτό μιλάμε για εις αξιολόγηση των κριτηρίων. Προσπαθήσαμε να, να έχουμε ε, μια σύσταση, αλλά τελικά αυτό το οποίο απεδείχθη είναι ότι απαιτείται μια δεσμευτική, ένα ε, δεσμευτικό νομικό μέσο. Με τη νομική βάση που έχουμε, ε, μπορούμε να έχουμε όχι μόνο αμοιβαία αναγνώριση, αλλά και συντονισμό των απαραίτητων προϋποθέσεων Επιτρέπεται λοιπόν η συνθήκη στον νομοθέτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συντονίζει τις ε, προϋποθέσεις ε, για τα επαγγέλματα και να εκδίδει τις τα σχετικά νομικά μέσα. Γίνεται ε, εις βάθος εξέταση όλων των προϋποθέσεων, ούτως ώστε να, υπάρχει, να τηρείται η αναλογικότητα. Δεν παρεμβαίνουμε λοιπόν στις αρμοδιότητες των κρατών μελών, μόνο αξιολογούμε κατά πόσο ε, πρέπει να γίνεται ε, η ρύθμιση αυτή των νομικά κατοχυρωμένων ε, επαγγελμάτων με συγκεκριμένα, για συγκεκριμένα προσόντα και υπάρχει και η συμφωνία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου από την ομολογία του. Ο κατάλογος τον οποίο έχουμε είναι αρκετά μακρύς, αλλά είναι συμβατός με την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σε ορισμένε περιπτώσει μπορεί να μην είναι σχετικά τα κριτήρια, πάντω αυτά τα οποία έχουμε κρατήσει στο κατάλογό μα είναι ε, τα συγκεκριμένα κριτήρια που προκύπτουν από την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Είναι λοιπόν σίγουρα τα κριτήρια αυτά τα οποία έχουμε ε, επιλέξει δεν συμφωνώ με ε, την κριτική της κυρίας ε, Νίμπλε. Καταλαβαίνω ε, αυτά τα οποία είπατε, αλλά η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι αυτή για τη συγκεκριμένη πρόταση. η πρόταση περιγράφει ακριβώς τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να αξιολογείται με βάση την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Ευχαριστώ. Uh, Άλλα σχόλια. Α, ο κύριος Le Ναι, η συζήτηση αυτή είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, διότι παρατίθενται δύο διαφορετικές απόψεις που φαίνεται να είναι δύσκολο να συνδυαστούν. Η μία είναι της κυρίας Νίμπλερ και η άλλη της Κομισιόν. Πιστεύω πως θα πρέπει καλύτερα να λάβουμε υπόψη αυτή την αυτορύθμιση των ε, ε, επαγγελμάτων, γιατί όπως στη χώρα μου, τη Γαλλία, λειτουργεί αρκετά καλά τελικά. Και ίσως θα πρέπει να το διερευνήσουμε περισσότερο. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Σε κάθε περίπτωση σημειώστε παρακαλώ ότι η προθεσμία και υποβολή τροπολογιών είναι η 9η Μαΐου. Η μέρα της Ευρώπης. Στις 6 το απόγευμα. Okay. Uh, we continue... Μάλιστα. Συνεχίζουμε. Θα πρέπει να συνεχίσουμε. Το σημείο 19, όπου όμως έχει βασικά αναβληθεί. Αλλά πρέπει να σας διαβάσω κάτι, μια πληροφορία λόγω της απουσίας του εισηγητή. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η γραμματεία θα σας δώσει τώρα ένα έγγραφο της γραπτής γνωμοδότησης της Νομικής Υπηρεσίας του Συμβουλίου της 7 Δεκεμβρίου 2015 όσον αφορά τη δυνατότητα για τη στήριξη και ανάπτυξη νομικών ε, θέσεων. Έτσι λέγεται. Λόγω του ότι είναι επιστευτικό αυτό το έγγραφο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του Εσωτερικού Κανονισμού του Συμβουλίου, τα μέλη της Επιτροπής ε, Νομικών Υποθέσεων ε, έχουν προνομιακά πρόσβαση στο έγγραφο αυτό, αλλά σας παρακαλώ ε, παρακαλείστε μάλλον να μην το αποκαλύψετε στο ευρύ κοινό χωρίς προηγούμενη έγκριση. Επίσης μας ζητήθηκε να το μελετήσουμε και να το διατηρήσουμε μέσα εδώ στα γραφεία μας, στους χώρους ε, του Κοινοβουλίου και εν πάση περιπτώσει αν το βγάλουμε από το Κοινοβούλιο να το φυλάμε ως κόρονο φθαλμού. So please take note of that. Uh, and we... Οπότε παρακαλώ λάβετε το αυτό υπόψη και τώρα θα συνεχίσουμε με άλλα σημεία που είναι προσυζήτηση αλλά και κλεισμένων των θύρων. Οπότε όλοι όσοι δεν έχουν ε, εξουσιοδότηση για να συμμετέχουν σε μια συνεδρία και κλεισμένων των θυρών παρακαλώ να εξέλθουν ησύχως της αιθούσης.